την αντιμετώπιση του θέματος του φόρου κληρονομιάς ε, όσον αφορά τον κανονισμό μετά την έγκριση του κανονισμού από πλευράς της Επιτροπής ο κύριος Μπόγκ έχει τον λόγο παρακαλώ κύριε Επίτροπε έχετε τον λόγο Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την ρύθμιση για τα θέματα κληρονομιάς που εγκρίθηκε πέρυσι και τώρα αποτελεί μέρος της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετική νομοθεσία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κληρονομιάς δημιουργούσε προβλήματα σε σχέση με την χρήση των δικαιωμάτων από πλευράς εκείνων που κληρονομούσαν κάτι σε περίπτωση ε, ε, θανάτου και εδώ τα συγκεκριμένα ωφέλη όσον αφορά τις διατάξεις μιας απλουστευμένης διαδικασίας οδηγούν σε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Αυτό το νομοθέτημα είναι ένα από πολλά παραδείγματα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να επιλύσει καθημερινά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και να εξοικονομήσει και κονδύλια. Και η ρύθμιση όπως για οποιοδήποτε νομοθέτημα που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ τελείως διαφορετικών εθνικών νομικών συστημάτων μπορεί να δημιουργήσει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής, υλοποίησης στις καθημερινές πρακτικές, στην καθημερινή πρακτική. Για την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε τέτοιων αναφιόμενων προβλημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί αρκετά χρόνια προωθούσε σχέδια τα οποία θα ευνοούσαν τους πολίτες να βρουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, της διασύνδεσης των μητρώων όσον αφορά διαθήκες σε σχέση με τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν διευκολύνσεις πανευρωπαϊκά. Ένα από τα πρώτα θέματα είναι, για παράδειγμα, ε, η ρύθμιση της, ε, ε, του θέματος της διαθήκης. Ο εντοπισμός της διαθήκης είναι ένα κέριο στοιχείο για την ε, κίνηση αυτής της διεργασίας. Ένα διαφανές σύστημα ανταλλαγής ε, πληροφοριών είναι ένα άλλο σχέδιο για τα θέματα κληρονομιάς ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εύληπτο, εύληπτα θέματα για τους πολίτες, ώστε στην ιστοσελίδα Succession in Europe, η κληρονομιά στην Ευρώπη, να μπορεί να αποτελεί στοιχείο άντλησης, πηγή άντλησης στοιχείων για τους πολίτες. Μία ρύθμιση που θα διευκολύνει τα πράγματα. Πέρυσι ένα εκατομμύριο ευρώ δώσαμε για δράσεις όσον αφορά το Συμβούλιο Συμβολεογράφων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση 14 εγχειρημάτων δράσεων κατάρτισης ώστε να καταρτιστούν συμβολεογράφοι πανευρωπαϊκά. Επίσης εργαζόμαστε για την δημιουργία της ε, επίλυσης προβλημάτων ε, σε θέματα διαθήκης και κληρονομιάς. Και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση EJN ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση πληροφοριών όσον αφορά τις εθνικές νομοθεσίες και διαδικασίες ε, για τα ευρωπαϊκά ε, νομοθετικά θέματα. Και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε μια μελέτη για να εξεταστεί η ανάγκη να ε, υπάρξουν μητρώα τέτοιων διαθήκων για την διευθέτηση θεμάτων κληρονομιάς και να υπάρχει διαλειτουργικότητα που θα διασφαλίζεται μεταξύ αυτών των συστημάτων σε σχέση με τα διαφορετικά διαφορετικά κράτη-μέλη. Δεν αφορά όμως την φορολογία αυτή η ρύθμιση που εδώ θα πρέπει να αξιολογείται πώς θα πρέπει να ρυθμίζεται και είναι διαφορετικό θέμα ε, πανευρωπαϊκά. Και μόνο ένα σε σχέση μετά την ε, ρύθμιση ε, όσον αφορά διπλάς, διπλή ή πολλές φορές και τριπλή φορολογία καταλήγουν στο να απολάβουν αυτά τα χρήμα, αυτού, αυτούς τους πόρους οι, όσοι έχουν δικαίωμα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε γιατί αρκετά κράτη έχουν, επιβάλλουν φορολογία για επί της ίδιας ε, ε, κληρονομιάς ε, ή επιβάλλουν μεγαλύτερη φορολογία επί συγκεκριμένης κληρονομιάς. Παρακαλώ να επιβραδύνετε παρακαλεί ο Πρόεδρος στον ομιλητή. Ο, η συνολική αξία λοιπόν μιας διασυνοριακής τέτοιας υπόθεσης μπορεί να πρέπει να πληρώνεται και όσον αφορά τους ε, ε, φόρους που πρέπει να καλυφθούν και επειδή αρκετά κράτη μπορεί να διεκδικούν το δικαίωμα φορολόγησης της ιδίας κληρονομιάς ή φορολογούν τους αλλοδαπούς κληρονόμους περισσότερο από ότι τους ε, γηγενείς κληρονόμους. Σαν αποτέλεσμα, πολίτες μπορεί να αναγκάζονται να πολλούν ιδιοκτησία τους για να καλυφθούν τα φορολογικά χρέη. Και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τα όσον αφορά ε, την κληρονομιά τους. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ε, προσκόμματα και εμπόδια, τα οποία θα παρακολύουν ίσως τους Ευρωπαίους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους διασυνοριακά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την φορολογία μπορεί να είναι ένα τεχνητό αντικίνητρο όσον αφορά την πρόθεση της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε κατά τα άλλα βιώσιμες επιχειρήσεις. Ε, λόγω του φόβου υπερβολικής φορολογίας και ε, λογαριασμών που θα έπρεπε να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες ε, θα μπορούσαν να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά για παράδειγμα την ρευστοποίηση ή την απόσυρση από τις επενδύσεις αυτές διασυνοριακά και όλα αυτά επειδή μπορεί να μην βλέπουν να υπάρχει πρόσθετη αξία στο να διατηρείται ένα, ε, ένα τέτοιο υψηλά φορολογήσιμο επίπεδο επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου 2011 υιοθέτησε μια ε, οδηγία, πώς, ε, μια σύσταση, πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποφύγουν διπλή φορολόγηση τέτοιου είδους κληροδοτημάτων. Ταυτόχρονα έδωσε και κατευθυντήριες γραμμές προς ανατολισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη πώς να διασφαλίζουν ότι διασυνοριακά τέτοιοι κανόνες όσον, αφορούν, όσον αφορά την φορολόγηση δεν θα συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση. Ο στόχος είναι απλούστατος. Το να δραστηριοποιηθούμε, να αντιμετωπιστεί το ε, θέμα των προσκομμάτων φορολογικά σε περιπτώσεις κληρονομιών διασυνοριακά και η επίλυση προβλημάτων διπλής φορολογίας. Και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε με όλα αυτά ότι το συνολικό το επίπεδο φορολόγησης σε συγκεκριμένη κληρονομιά δεν θα είναι υψηλότερο από εκείνο της φορολόγησης που θα εφαρμοζόταν αν μόνο ένα κράτος μέλος είχε κυριαρχικά δικαιώματα να επιβάλλει φόρο σε αυτή την κληρονομιά και μόνο ένα αυτό ζητεί από τα κράτη-μέλη να ανακουφίσουν ε, φορολογικά ε, σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας τους ε, για φορολόγηση κληρονομιών και την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει έκθεση πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τα κράτη-μέλη και τις δράσεις τους για την αποφυγή διπλή διπλής φορολόγησης κατά το 2014. Αν η έκθεση αυτή του 2014 καταδείξει ότι διασυνοριακ... τα διασυνοριακά προβλήματα σε σχέση με την φορολόγηση εξακολουθούν να υφίστανται, τότε θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις στη διάθεσή της, ακόμα και την ανάγκη να αναλάβει νομική δράση ώστε να αρθούν, να εξαλειφθούν αυτά τα νομικά προσκόμματα. Εν τέλει, εν τω αυτή τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ευκαιρία να ζητήσει από όλα τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν και να εντείνουν τη συνεργασία του και να προχωρήσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστούμε θερμά. Πρώτο αγορητή, ο κύριος Τσβίφκα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, Κάνουμε λόγο απόψε εδώ για την ρύθμιση κληρονομικών δικαιωμάτων Σίγουρα είναι ένα κεκτημένο αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ότι φτάσαμε εδώ. Μεγάλη πολλή εργασία χρειάστηκε σε ένα σύνθετο περίπλοκο θέμα και υπήρχε και μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η σπουδαιότητα αυτή της ε, επίλυσης αυτών των προβλημάτων για τους πολίτες μας. Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν μια δυσχερή κατάσταση πολλές φορές διότι έχουν χάσει τους συγγενείς ή οικείους τους και βρίσκονται και σε μια κατά τα άλλα δυσχερή ε, νομική κατάσταση. Οι διατάξεις λοιπόν δίνουν στους πολίτες την δυνατότητα μέσω αυτών των διευθετήσεων να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, μια συγκεκριμένη νομολογία. Θα είναι σαφές ε, ποιες προϋποθέσεις ε, θα πρέπει να ισχύουν. Θα ήθελα όμως για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω κάτι εδώ. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις διατάξεις. Επ' αυτής της αρχής βασίζεται η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε νομικής διάταξης. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να προσθέσουμε κάτι εδώ. Το ότι το θέμα το ίδιο, το ζήτημα δηλαδή των κληρονομικών δικαιωμάτων σε περίπτωση τέτοιων κληρονομιών είναι πολύ περίπλοκο ακόμα και για νομομαθείς και νομικούς Κατά τούτο χρειάζονται ακόμα σαφέστερες λύσεις λοιπόν στις οποίες θα καταλήξουμε όσον αφορά το διεθνές πλαίσιο της διευθέτησης τέτοιων ε, κληρονομικών ε, ζητημάτων. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις λοιπόν και για να αντιμετωπιστεί η διπλή ή πολλαπλή φορολόγηση κιόλας. Διότι αυτή η διπλή, η διτή ε, φορολόγηση στον κανονισμό δεν ρυθμίζεται. <coughs> βλέπουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα για τους πολίτες όμως ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Επίτροπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι θέλετε να αντιμετωπίσετε και να εξαλείψετε αυτά τα προβλήματα. Αν οι διατάξεις ε, απλουστεύουν τα θέματα κληρονομιών τότε πρέπει να έχουν νομική βεβαιότητα οι πολίτες πώς θα εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ποιες συνέπειες και επιπτώσεις επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά, προτού ακόμα αρχίσουν να ισχύουν αυτά τα διεθνή δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ τον ε, κανονισμό για τις κληρονομικές διατοχές ένα από τα ωραιότερα επιτεύγματα αυτής της ε, θητείας. Μπορεί να φαίνεται μακρινό και δύσκολο το θέμα αυτό, όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει αγγίξει τους πολίτες την καθημερινή του ζωή ως Ευρωπαίους πολίτες. 450.000 είναι οι περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες κάποιες ε, οικογένειες κάθε χρόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν μια περίπτωση κληρονομικής διαδοχής και 120 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία συναλλάσσονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται υπαστοί μεταξύ δύο χωρών και οι οποίοι ε, πρέπει να βρουν λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματά τους. Εμείς λοιπόν καθορίσαμε ποιος είναι ο εφαρμοστέος νόμος σε αυτή την περίπτωση. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η συζήτηση την οποία εμείς ζητήσαμε και επί της οποίας άρχισε να δίνει κάποιες απαντήσεις ε, ο Επίτροπος. Γιατί εάν δεν απαντηθεί το φορολογικό πρόβλημα αυτό δηλαδή της διπλής φορολόγησης οπωσδήποτε θα υποστεί ζημία ε, αυτό το νομικό κείμενο. Γι αυτό, και εδώ ακριβώς ε, μπορώ να θυμηθώ αυτό που είπαμε και στη συζήτηση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Δηλαδή, ε, ε, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου θα πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά, βήμα βήμα, έτσι ώστε να δούμε πού ε, υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχει αδυναμία προώθησης των θεμάτων κλπ. Η διπλή φορολόγηση θα πρέπει να ξεπεραστεί το, η σύσταση του 2011 θα πρέπει να ε, υλοποιηθεί ουσιαστικά και αυτός ο νόμος θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα έτσι ώστε να έχει ε, καλή επίπτωση, θετική επίπτωση στην πραγματική ζωή των ε, πολιτών. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι τελευταίο. Με τον Ταντέους Φιέβγα, τη Σιζίλια Βίγκστρομ, που είναι συνάδελφοι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Βλέπετε, εμείς ε, δεν θέλουμε να μιλάνε οι εφημερίδες ε, για μας, ε, γιατί ο δικαστικός όπως και ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου είναι άτομο που πρέπει να εργάζεται στο, στη μοναξιά του έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό κάναμε και σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σεσίλια Βίκστρομ, επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν βλέπουμε ότι η έντολη αυτή έδωσε ευκαιρία να εργαστούν κάποιοι σκληρά για μια νομική ρύθμιση αυτού του θέματος και είμαι πεισμένη ότι οι διασυνοριακές, τα θέματα διασυνοριακών ε, κληρονομικών ε, διαδοχών και δικαιωμάτων θα μπορέσουν να διευθετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ότι δίνεται συνέχεια σε αυτά τα θέματα και εξετάζεται η φορολόγηση σε ποια χώρα θα επιβάλλεται όταν έχουμε διάφορες υποψήφιες χώρες ε, για επιβολή τέτοιας φορολόγησης. Ε, και έχουμε πολίτες που αντιμετωπίζουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση, έχουν τελείως διαφορετική πληροφόρηση και στοιχεία, αν κάποιο ακίνητο για παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο κληρονομούν και τα θέματα τα φορολογικά εντάσσονται στις αρμοδιότητες των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ αυτά τα συστήματα είναι τα αρμόδια. Δεν είναι όμως εύθετο η πολίτες να υποβάλλονται σε διτή, διπλή φορολόγηση όταν έχουν ένα τέτοιο κληροδότημα το οποίο ε, διεκδικούν να φορολογήσουν ε, περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. Και εδώ θα πρέπει να ρυθμιστούν τα θέματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι κανόνες να είναι εύληπτοι, να είναι απλοί και να μην είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να καταβάλουν διπλό φόρο. Θα ήθελα να γνωρίζω κύριε Επίτροπε ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία έχετε ακολουθήσει και αναλαμβάνετε ώστε να απλουστευτούν και να διευκολυνθούν αυτά τα θέματα. Θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να υπάρξει σαφήνεια για τους πολίτες. Θα προχωρήσουμε σε αυτά ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Μπόντο, συνάδελφος Μπόντου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, πρόσφατα η κινητικότητα των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ε, προβλήματα ε, για τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές. Νομίζω ότι η ιδιοκτησία προκαλεί, η κυριότητα προκαλεί την εφαρμογή πολλών νομοθεσιών κληρονομιάς και δημιουργεί συγκρούσεις νόμων ε, το κανονισμό των ε, κληρονομικών διαδοχών σε περιλαμβάνει την αρχή ότι ένας νόμος, ένα δίκαιο πρέπει να εφαρμόζει ε, προσδιορίζοντας τον τόπο διαμονής του θανόντος. Ε, προηγουμένως δεν υπήρχε προγραμματισμός ε, για την φορολόγηση. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 έχουμε τη σύσταση της Επιτροπής ε, για να αποφευθεί η διπλή φορολόγηση των κληρονομιών και έχουμε την έκθεση του 2000, θα έχουμε την έκθεση του 2014 να δούμε ποια θα είναι η λύση. Θα υπάρχει ίσως ένα πιστοποιητικό για την αποφυγή της διπλής ε, φορολογίας, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα των κληρονομικών διαδοχών. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία συνάδελφος Ρέγνερ έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Με τον κανονισμό και ρύθμιση αυτών των θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα κληρονομιών η ζωή πολλών πολιτών μπορεί να βελτιωθεί. Όταν έχουμε τώρα το θέμα της διπλής φορολόγησης φυσικά είναι και κοινωνικά τεράστια σημασία. 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, γυναίκες και άνδρες αφορώνται άμεσα από αυτό σε σχέση με όσους ε, διαμένουν εκτός της ε, χώρας τους. Και έτσι, σε σχέση με κληρονομικά δικαιώματα, θα πρέπει να επιλέγουν τι θα συμβαίνει σε σχέση με την τελευταία έδρα στην οποία, την οποία είχαν ε, προτού λόγω της αποβίωσης ε, και της ε, ε, διαθήκης θα πρέπει να ρυθμιστούν θέματα φορολογίας. Θα πρέπει να αποφύγουμε χρονοβόρες διαδικασίες όπως και διπλή φορολόγηση και πρέπει να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κενά και χάσματα που υπάρχουν. Και εδώ εν δυνάμει θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους κοπέλους. Αν φοβάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοιου είδους φορολογική επιβάρηση θα αφορά πολλούς πολίτες ε, που θα ε, έχουν το πρόβλημα της ε, καταβολής της, των φόρων στις αρμόδιες εφορίες. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει ακριβώς να τα αντιμετωπίσουμε και να αποφύγουμε να δημιουργούνται προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία. Και μέσα, μέσω της διαδικασίας Catch the Eye η κυρία Μπασέσκου είναι εκείνη που θα παρέμβει παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα ποιο είναι σε σχέση με τα πιστοποιητικά ε, τις διαθήκες ε, επιλήθηκε σε σχέση με μια ρύθμιση του 2012. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με τη διαφορετική φορολόγηση που υφίστανται κληροδοτήματα ή μάλιστα και της απλά επιβαλόμενης πολλαπλής φορολόγησης και θα πρέπει εδώ σε σχέση με τα προβλήματα αυτά στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου είμαι αντιπρόεδρος να εξετάζονται ε, ε, ε, σε βάθος. Με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό κληρονομιάς διευθέτησης των θεμάτων κληρονομικής διαδοχής ε, πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα τελεσίδικα και όχι με μια ε, σύσταση για αποφυγή διπλής φορολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Θα δημιουργούσαμε επίσης ένα χώρο για την ε, ασφάλεια και την ελευθερία και δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και με την παρέμβαση του κυρίου Μποργκ Κλίνη. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήταν ο Βεριαμίν Φρανκλίνος εκείνος, ο οποίος το 1789 είπε ότι Τίποτα στη ζωή δεν είναι βεβαιότερο από τον θάνατο και τους φόρους. Και εδώ ακριβώς ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα ε, της ε, κληρονομικής διαδοχής και όσον αφορά και τα θέματα τα φορολογικά. Θα ήθελα να απαντήσω το ερώτημα το οποίο διατυπώθηκε προηγούμενα από προλαλήσασα για το ποιο κράτος είναι εκείνο το οποίο θα επιβάλλει φορολογία και θα εισπράττει φόρους επί Δεν αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την ε, πρόταση αυτή αυτό το ζήτημα, εκτός από το ότι λέμε ότι το συνολικό ποσό του φόρου κληρονομιάς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το οποίο θα ήταν φόρος κληρονομιάς αν μόνο ένα μόνο και μόνο ένα κράτος μέλος ήταν υπεύθυνο και αρμόδιο να επιβάλλει ε, φόρο από πλευράς του και μόνο. Αυτό λοιπόν ε, λέμε και ότι σε σχέση με την φορολόγηση στόχος πρέπει να είναι να πετύχουμε ότι το συνολικό επίπεδο φορολόγησης επί μια συγκεκριμένης ε, συνολικά κληρονομιάς δεν θα είναι ποτέ υψηλότερο από το επίπεδο εκείνο το οποίο θα ίσχυε και θα επεβάλλεται αν μόνο ένα κράτος μέλος αποκλειστικά είχε φορολογικά κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία θα ζητούσε να καλυφθούν σε σχέση με μια τέτοια κληρονομική διαδοχή. Αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια, ότι δεδομένου του συνολικού φόρου που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτή την φορολόγηση από ένα κράτος και μόνο αν αυτό επέβαλε από πλευράς του τον φόρο, θα μπορούσε και να συλλεγεί το ποσό αυτό και από τρία διαφορετικά κράτη-μέλη. Δεν επεμβαίνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ε, ρυθμίζουμε εμείς το πόσα κράτη-μέλη θα επεμβαίνουν και θα εισπράττουν φόρους. Όμως το συνολικό ε, ποσό το οποίο θα επιβάλλεται δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον φόρο που θα επέβαλε ένα και μόνο κράτος μέλος επί μιας τέτοιας κληρονομικής διαδοχής. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές και όταν συνδέονται αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή το θέμα της κληρονομιάς και το, της φορολόγησης, βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος ε, προβλημάτων με, τις, ε, την πολλαπλή φορολόγηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της διασυνοριακής φορολόγησης μπορεί να είναι πραγματικά θέμα το οποίο θα κολλεί και θα επιβαρύνει τους πολίτες. Λοιπόν, μικρές αλλαγές στις διατάξεις από πλευρά των κρατών μελών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγματικά ωφέλη για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σχέδιο και εγχείρημα τώρα είναι και πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε και να δούμε πώς αυτή η σύσταση θα εφαρμοστεί και θα υλοποιηθεί στα διάφορα κράτη-μέλη και έχω και εντολή από πλευρά της Επιτρόπου Ρέντινγκ να δηλώσω ότι αν τα αποτελέσματα αυτή τη σύσταση δεν υλοποιούνται με ικανοποιητικό τρόπο, τότε θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια δεύτερη φάση ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλοντας, καταθέτοντας νομοθετικές προτάσεις. Και αυτό θα ωφελούσε πάλι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ελπίζω ότι ε, αρχές στα κράτη-μέλη σε σχέση με το έτος αυτό το οποίο θα μεσολαβήσει θα σημειώσουν προόδους ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και ολοκληρώνεται έτσι εδώ η συζήτηση επ' αυτού του θέματος της ημερήσιας διάταξης απόψε και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της απόψινής μας συνεδρίασης που είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού υπαριθμών 1049 κάθετος 2001. Και θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο.